Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής, υπάτηση εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, με θέμα η κατάσταση στη Γεωργία. Ε, εξ ονόματος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και υπάτηση εκπροσώπου, το λόγο έχει ο κύριος Μαυρογιάννης Ανδρέας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να πάρω το λόγο στην αρχή της συζήτησης αυτής εξ ονόματος της υπάρχης εκπροσώπου της κυρίας Άστον. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του τη 17η Νοεμβρίου του 2011 στήριξε την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας και την διαδικασία δημιουργίας πολιτικής και εταιρικής σχέσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία της Γεωργίας. Αναγνώρισε επίσης τη σημασία της διαδικασίας της Γενέβης και στήριξε τις ε, ενέργειες του ειδικού αντιπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Νότιο Κάφκασο και της Επιτροπής Παρακολούθησης της Κατάστασης. Τα μέλη του σώματος, του σώματος αυτού υποστήριξαν και τις προσπάθειες για την εμβάθυνση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γεωργία. Στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Euronest στον Μπακού τον Απρίλιο, έγινε δεκτό ένα ψήφισμα το οποίο υπογραμμίζει τη σημασία της ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών, της ενίσχυσης της δημοκρατίας της ε, ε, ελευθερίας ε, της πολιτικής δραστηριότητας, της ελευθερίας του τύπου και επιπλέον αυτού πολλά μέλη έχουν υποβάλει κοινοβουλευτικές ερωτήσεις σχετικά με την αντιμετώπιση της αντιπολίτευσης, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών σχέσεων και άλλων σχετικών θεμάτων. Όλα τα θέματα αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία γιατί εμείς παρακολουθούμε την προετοιμασία των εκλογών το φθινόπωρο και υποστηρίζουμε τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της Γεωργίας οι οποίες εδράζονται στην αρχή της συνένεσης. Ο κ. Ρομπάι ο πρόεδρος Ρομπάι είναι στη Γεωργία σήμερα. Η επίσκεψή του είναι ευκαιρία να αποδείξει το υψηλότερο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις σχέσεις μας με την Γεωργία και στην ειρηνική εξέλιξη του συνόλου της περιοχής του Νοτιού Καυκάσου. Εγώ δεν θα προκαταλάβω τα μηνύματα του Προέδρου Βαν Ρομπάη προς τους Γεωργιανούς σήμερα, αλλά παρόλα αυτά θα ήθελα να υπογραμμίσω ορισμένα πολύ σημαντικά για μας θέματα, πριν ξεκινήσει η συζήτηση. Έχουμε επιτελέσει σημαντικά βήματα με τη Συμφωνία Σύνδεσης και στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για μια εμπορική σχέση, εταιρική σχέση, ένα πρόγραμμα δράσης μέτρων το οποίο θα επιτρέψει την κινητικότητα και θα ενισχύσει τις επαφές ανάμεσα στις δύο, στους δύο εταίρους αλλά για να προχωρήσει η διαδικασία είναι απαραίτητο η Γεωργία να κάνει τα απαιτούμενα βήματα στο πνεύμα ακριβώς των ρυθμίσεων της Συμφωνίας Σύνδεσης. Εμείς στηρίζουμε τη Γεωργία σε όλα τα επίπεδα, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες που έχει να εφαρμόσει την αρχή ε, more for more στα αγγλικά. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν ο πρόεδρος Μπαρόσο, ο επίτροπος Φίλε και η αντιπρόεδρος Άστον έχουν ε, υπογραμμίσει προς τον πρόεδρο Φίλη στην τελευταία τους πρόσφατη συνάντηση στις Βρυξέλλες την ανάγκη που υπάρχει να διασφαλιστεί ο δίκαιος πολιτικός ανταγωνισμός και η νομιμοποίηση των εκλογών. Οι εκλογές τον Οκτώβριο, οι κοινοβουλευτικές εκλογές θα πρέπει να είναι στο επίπεδο των διεθνών δημοκρατικών προτύπων και η εμπιστοσύνη ε, της κοινή γνώμης είναι ε, καθοριστική για μας. Θα πρέπει να υπάρξει μια αξιόπιστη και ισχυρή αντιπολίτευση η οποία να συμμετέχει στις εκλογικές διαδικασίες ε, σεβόμενοι φυσικά τη συνταγματική τάξη και τον νόμο. Έχουμε την αίσθηση ότι εν μέρει η κυβέρνηση προσπαθεί να παρεμποδίσει τη συμμετοχή του ηγέτη της αντιπολίτευσης ε, στη διαδικασία του Ιβάν Νισβίλη. Και ότι ο νόμος εφαρμόζεται μονομερός θα πρέπει να επιμείνουμε έτσι ώστε οι νομικές προβλέψεις να εφαρμόζονται με πολύ δίκαιο τρόπο, αντικειμενικό τρόπο, έτσι ώστε να μην υπάρξει αμφιβολία για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η, η προεκλογική εκστρατεία. Επίσης παρακολουθούμε από κοντά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί την οικονομική του επιφάνεια ο ηγέτης της αντιπολίτευσης ε, για εκλογικούς λόγους, για εκλογικά κέρδη. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να παρακολουθήσουμε προσεκτικά γιατί η ψήφος δεν αγοράζεται και θα πρέπει επίσης να υπάρχει η ισομερής πρόσβαση και στα μέσα ενημέρωσης γιατί από ό,τι φαίνεται τα δύο δημόσια, τα δύο δημόσια κανάλια στην Γεωργία έχουν ε, ε, επιμείνει προς την κατεύθυνση αυτή περισσότερο από τα ιδιωτικά. Σημειώνουμε επίσης και τις δηλώσεις του Προέδρου γύρω από τα θέματα αυτά, αν και θα θέλαμε βέβαια την εφαρμογή όλων αυτών των κανόνων ισοτιμίας να τα συζητήσουμε περισσότερο. Να υπογραμμίσω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπέρ πάντα της επίλυσης των διαφορών, των συγκρούσεων, των προσπαθειών που γίνονται στη Γεωργία υποστηρίζοντας φυσικά πάντα την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας, συνεισφέροντας στη σταθερότητα της χώρας αυτής μέσω της, επιστολή, της αποστολής ε, παρατήρησης και συμμετέχοντας στην διαδικασία των συζητήσεων στη Γενέβη. Το πρόβλημα της Απχαζίας και της Νότιας Οσετίας είναι κάτι το οποίο παραμένει πολύ σημαντικό για μας και θα κάνουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση. Η προσπάθειά μας αυτή φαίνεται και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 27 Φεβρουαρίου 2012. Προσβλέπω στις, στο να ακούσω πολύ προσεκτικά και να λάβω υπόψη μου τις απόψεις των αγαπητών μελών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από της Προεδρίας, ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων, εξ του ΕΛΚ, το λόγο έχει ο συνάδελφος κύριος Λίσεκ για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι. Είμαι σε θέση να εργαστώ επί 1,5 χρόνο για την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ε, Συμφωνία Εταιρική Σχέση ΕΕ και Γεωργίας. Επισκέφθηκα αρκετές φορές ε, την Γεωργία και είχα πάνω από 10 συναντήσεις και με την αντιπολίτευση και με εκπροσώπους της κυβέρνησης και με τον Ομπουσμαν ε, ε, και τα μέσα και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και με εκείνους ε, που συνεργάζονται με την κυβέρνηση και με εκείνους που συνεργάζονται με την αντιπολίτευση και την κοινοβουλευτική αλλά και την εξωκοινοβουλευτική αντιπολίτευση. Θα ήθελα να παρουσιάσω τις απόψεις μου επ' αυτού του θέματος. Προτού το κάνω αυτό θα ήθελα αν επιτρέπετε να σας υπενθυμίσω το ψήφισμά μας, δύο εδάφια αυτού του ψηφίσματος που με 90% των ψήφων του Ευρωκοινοβουλίου εγκρίθηκε. Αναφέρουμε ότι θα έπρεπε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για την δημοκρατική πρόοδο που έχει επιτευχθεί από πλευρά της Γεωργίας στην παγίωση των ε, δημοκρατικών θεσμικών οργάνων όπως του συνηγόρου, του ομπουτσμάν, ε, του δικαστικού συστήματος και των οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Θα έπρεπε, προσθέτουμε, να συγχαρούμε την Γεωργία για τα χαμηλά ποσοστά, χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητα. Σε ένα άλλο σημείο λέμε ότι θα θέλαμε να ζητήσουμε από την κυβέρνηση της ε, Γεωργίας να προβεί σε ε, επικοδομητικό διάλογο με την αντιπολίτευση και να προωθήσει ε, μέτρα εκδημοκρατισμού υπέρ τη ελευθερία έκφραση. έκφρασης. ομιλείτε γρήγορα πολύ, λίγο πιο αργά. <laughs> Σας ευχαριστώ πολύ για την παρατήρησή σας, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να ακολουθήσω βραδύτερο ρυθμό. Λοιπόν, συνεχίζω. Σήμερα νομίζω ότι όλοι όσοι υπερψηφίσαμε αυτά τα εδάφια, αυτό το ψήφισμα και επενέθηκε η Γεωργία όχι μόνο από εμάς ε, πολιτικούς άνδρες αλλά και από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, από την ε, Transparency International ε, για τον εκδημοκρατισμό και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Οι τελευταίες εκλογές υπέρ των εκπροσώπων των δημοτικών αρχών θετικά σχολιάστηκαν από τους παρατηρητές. Ακόμα και αντιπολίτευση ανέφερε ότι δεν υπήρχε υπήρξαν και ότι διασφαλίστηκαν οι διεθνείς προδιαγραφές κατά τις εκλογές αυτές. Επανέρχομαι στα θέματα που είναι υποσυζήτηση. Τι συνέβη ώστε να πρέπει να ξανασυζητήσουμε τα θέματα της Γεωργίας ακόμα μία φορά. Νομίζω ένα μείζον γεγονό ε, συνέβη και αναφέρθηκε από τον Υπουργό. Έχουμε ένα νέο σώμα, ένα νέο φορέα, ένα νέο ηγέτη της αντιπολίτευσης ε, που ανεφεί, κάποιον που είναι δισεκατομμυριούχος, έχει δισεκατομμύρια δολάρια, έχει περισσότερα χρήματα από ότι ο εθνικός προϋπολογισμός της ίδιας της Γεωργίας ως κρατικής οντότητας. Όμως αυτά τα χρήματα δεν τη χάνουν καλής ε, χρήσης. Θα μπορούσα να μιλήσω από προσωπικά βιώματα που είχα κατά τους τελευταίους μήνες, αλλά όλοι έχουμε και αντίστοιχα βιώματα. Επί αρκετούς μήνες τώρα είδαμε κάποιες πληροφορίες ε, που ε, έρχονται από την Γεωργία ότι ο πρόεδρος λέει Σακασβίλη είναι τέρας και για τα όσα συμβαίνουν και τεκταίνονται από το ε, κόμμα, το ε, κυβερνητικό κόμμα και πώς παραβιάζεται το κράτος δικαίου, ε, οι νόμοι κτλ. Αποφάσισα να διακριβώσω αυτά τα θέματα και να δω τι συμβαίνει και φαίνεται ότι μια ομάδα γερμανικών και βρετανικών αρχών μίσθωσαν ένα άτομο για να εργαστεί υπέρ αυτών των συμφερόντων του. Και θέλω να τονίσω ένα πράγμα με ιδιαίτερη σαφήνεια. Η ύπαρξη τέτοιων ε, μηνυμάτων και τέτοιων προσπαθειών δεν στέφεται ποτέ με επιτυχία. Αυτό θα ήθελα να αναφέρω. Ευχαριστώ. Ρούτσεκ για λεπτό. Ευχαριστώ. Όπως είπε ο κύριος Μαυρογιάννης προηγουμένως, ο πρόεδρος Φαν Ρομπόι είναι στην Γεωργία. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ο επίτροπος Φιούλε στην ε, Γεωργία. Αυτό δείχνει τη σημασία που αποδίνουμε στη χώρα αυτή και τη συνόλη περιοχή. Είναι λοιπόν επιθυμία μας και όλων των σοσιαλδημοκρατών η Γεωργία να επιτύχει στο εγχείρημα αυτό στις πολιτικές μεταρρυθμίσεις, στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, να καταφέρει να διατηρήσει την εδαφική της ακαιρεότητα και φυσικά να ευδοκιμήσουν και οι διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης <clears throat> Γεωργίας και έτσι να επιτευχθεί ταχεία πρόοδος στο διάλογο για την φιλελευθεροποίηση των προξενικών θεωρήσεων. Με στόχο φυσικά να υπάρξει απαλλαγή για τους κατοίκους Γεωργίας από την υποχρέωση βίζας. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ θετικά και θέλουμε να χαιρετήσουμε τις ε, μεταρρυθμίσεις που επετέφθησαν τους τελευταίους μήνες και τα τελευταία χρόνια στην Γεωργία. Όπως ξέρουμε όμως θα έχουμε κοινοβουλευτικές και προεδρικές εκλογές πολύ σύντομα στη Γεωργία και βλέπουμε ότι υπάρχουν σημαντικές εντάσεις στη Γεωργία και ανεβαίνει το θερμόμετρο. Επομένως, οι φίλοι μας στη Γεωργία και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση θα πρέπει να καταπραίνουν τα πνεύματα. Χρειάζονται αδιάβλητες και ελεύθερες εκλογές η Γεωργία. Χρειάζονται σωστές προεκλογικές εκστρατείες όπου όλα τα πολιτικά κόμματα, όλες οι πολιτικές παρατάξεις και η αντιπολιτευτική, ο αντιπολιτευτικός συνασπισμός να έχουν πλήρη πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης. Θα είναι κέρυες αυτές οι εκλογές τόσο για τη Γεωργία είναι σημαντικό να διατηρήσουμε λοιπόν τον ανοιχτό χαρακτήρα και το αδιάβλητο των εκλογών και προσδοκούμε όλοι στο να υπάρξει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία σύνδεση και τη φιλελευθερωποίηση στι προξενικές θεωρίε. Εξ ονόματο των Σοσιαλδημοκρατών λοιπόν θέλω να ευχηθώ κάθε επιτυχία στου φίλου μας από τη Γεωργία. Τώρα εξ ονόματο της ομάδος Άλντε το λόγο έχει η συνάδελφο κυρία Νόρικα Νικολάη για δύο, λεπτό. δύο λεπτά. Uh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος της ομάδας των φιλελευθέρων θα ήθελα να τονίσω ότι εμείς υποστηρίζουμε, όπως έχουμε και στο παρελθόν πάντα υποστηρίξουμε, μια δημοκρατική γεωργία. Μια γεωργία ευημερούσα η οποία θα μπορούσε έτσι να εξασφαλίσει την επίτευξη των ευρωπαϊκών προτύπων και προδιαγραφών. Πιστεύω ότι σημαίνει συζήτηση είναι μια συζήτηση μεταξύ της εξουσίας και της αντιπολίτευσης, της αριστεράς και της δεξιάς. Αν κάποιος βρίσκεται στην εξουσία δεν πρέπει να ανησυχεί για, τα, για τη θέση της αντιπολίτευσης. Αλλά ο πρόεδρος Σακιασβίλη για πρώτη φορά ανησυχεί για το γεγονός ότι είναι ισχυρή και ενωμένη η αντιπολίτευση στην Γεωργία. Φυσικά υπάρχουν καταγγελίες που εκτοξεύονται από τη μία πλευρά έναντι της άλλης. Ε, οι κατηγορίες αυτές, οι καταγγελίες αυτές δεν έχουν φυσικά αποδεχτεί. Για μένα η δημοκρατία δεν είναι ένας ανοιχτός πόλεμος μεταξύ των τηλεοπτικών καναλιών που ανήκουν στην κυβέρνηση στην αντιπολίτευση. Δεν είναι ένας πόλεμος στα μύρια. Βλέπουμε λοιπόν όλο και περισσότερες τηλεοπτικές ε, ε, τηλεοπτικά κανάλια να αναλώνονται μόνο στα θέματα αυτά. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να υπάρξει η επιζήτηση ενός μονοπωλίου για την αλήθεια, κάτι το οποίο διαφρώνει και τη δημοκρατία μια τέτοια προσπάθεια. Κατά την άποψή μου λοιπόν, η κατηγορία ότι ένα κόμμα παραδείγματος έχει στην ε, ε, κεφαλή του ένα άτομο με μεγάλη οικονομική επιφάνεια δεν σημαίνει τίποτα ο πλούτος και η ένδια δεν είναι από μόνες τους αρετές ή κακίες μπορούν να δημιουργήσουν ίσως κάποιες αμφιβολίες για την αξία των ατόμων που έχουν ή δεν έχουν αυτή την περιουσία. Αλλά θα πρέπει να έχουμε μια συζήτηση η οποία βασίζεται σε ιδέες, σε οράματα και σε προγραμματικές απόψεις, όχι μια παράλληλη συζήτηση η οποία ουσιαστικά καθοδηγείται από τα κόμματα και τα μεσαριμένες. Το είπε και ο Επίτροπος Φιούλε. Αυτές οι εντάσεις που επισκιάζουν την προεκλογική διαδικασία της Γεωργίας μπορεί να αποβούν πολύ επικίνδυνες στο μέλλον. Η τωρινή κυβέρνηση λοιπόν θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι εκλογέ θα γίνουν μέσα σε ένα γαλήνιο κλίμα και μέσα στα πλαίσια των δημοκρατικών κανόνων και προδιαγραφών. Μόνο με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι η Γεωργία θα έχει ένα ελεύθερο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. ομάδα των Πρασίνων είναι η συνάδελφος κυρία Ούλρικε Λούνατσεκ, ομοίω για δύο λεπτά. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω πως η συζήτηση που έχουμε δείχνει ακριβώς γιατί χρειάζεται μια τέτοια συζήτηση. Γιατί είχαμε και επίσκεψη εδώ πέρα πολλών Γεωργιανών από την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση, τη νέα Ηνωμένη Αντιπολίτευση ε, ακούμε πολλά και διάφορα και δεν είμαστε εμείς βέβαια αυτοί που θα πάρουμε το πλευρό του ενός ή του άλλου. Εμείς θα ορίσουμε αυτό το οποίο ε, πρέπει να κάνει μια σύγχρονη δημοκρατική χώρα. Αυτό ε, για το οποίο ανησυχώ είναι πως ε, δεν ξέρω αν θα πρέπει εμείς να προειδοποιήσουμε πολίτες, κυβέρνηση αντιπολίτευση για τη Γεωργία. Πώς ο πόλεμος των λέξεων και οι αδιαφανείς εκλογές είναι κάτι το οποίο βλάπτει το, την εικόνα της Γεωργίας, όχι του Κωσυφοπεδίου, όχι μόνο στο Κοινοβούλιο αλλά στην Ευρώπη. Και να διαβάσω μια δήλωση, αν μου επιτρέπετε, του Ινστιτούτου Δημοκρατίας που λέει πως ανησυχεί για την πόλωση στη χώρα και την έλλειψη πολιτικής κουλτούρας μεταξύ των πολιτικών ηγετών. Οπότε πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως ε, ο πόλεμος ε, των λέξεων δεν είναι κάτι το θετικό. Χρειάζεται επίσης διαφάνεια της χρηματοδότησης των κομμάτων. Για όλους. Κυβέρνηση, αντιπολίτευση. Και εμένα δεν μου αρέσουν οι ολιγάρχες ε, στην πολιτική, αλλά το πόσα λεφτά έχει κανείς δεν πρέπει να είναι κριτήριο του εάν θα εκλέγεται ή όχι. Όπως είπε και η προηγούμενη ομιλήτρια, το θέμα είναι οι ιδέες και η θέληση να βελτιώσει κανείς ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και όλα αυτά στη χώρα. Θετικό ήταν για τα ΜΜΕ πως ε, κάθε καλωδιακό δίκτυο πρέπει να μεταδώσει ε, τα μηνύματα των πολιτικών κομμάτων. Κάτι το οποίο με ενισχύει είναι πως είναι πολύ γεμάτες φυλακές στη χώρα. Ναι, έπεσε ε, η εγκληματικότητα, αλλά για κάποιοι ακτιβιστές, για μικροπράγματα, έτσι, χουλιγανισμό, καταδικάστηκαν σε 35 μέρες φυλακής. Κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει σε προεκλογική περίοδο. Ε, και καλό κυβέρνηση, αντιπολίτευση να ηρεμήσουν λίγο και να έχουμε ελεύθερες και δίκες εκλογές. Λούνατσεκ, κύριε Λίσεκ, θέλεις να κάνετε χρήση της μπλε κάρτας. Excuse me, it's me. Τόμας Χορέντα. Εγώ είμαι ο Τόμας Χορέντα. Okay. Ah, okay. Thank you. Ε, Πήγα στη Γεωργία με την κυρία Νικολάη μαζί. Κυρία Νικολάη, δεν σας είδαμε πριν, τώρα έχουμε, υπάρχει επόμενη ομιλητής. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ε, επόμενος ομιλητής εξ, ονόματο ECR είναι ο συνάδελφο κυρίως Πορέμπα. Για ένα λεπτό. Panie Przewodniczący, Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, επί μακρόν διερωτώμην γιατί συζητούμε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό το θέμα. Πρόσφατα πέρασε μια καλή έκθεση εδώ του κυρίου Λίσεκ όπου επενήσαμε την συνέπεια των εφαρμογών των δημοκρατικών προτύπων στη Γεωργία και έκτοτε διερωτώμε τι συνέβη. Τίποτα δεν συνέβη έκτοτε. Αντιθέτω, οι αρχέ τη Γεωργία εξακολουθούν να κάνουν μεταρρυθμίσει εφαρμόζουν τις, τα διάφορα ευρωπαϊκά, τα δημοκρατικά πρότυπα, εφαρμόσαν το νέο νόμο για τα μέσα ενημέρωσης, μεταρρύθμισαν τον εκλογικό νόμο και όσον αφορά το εμπόριο είναι πολύ υψηλά όσον αφορά το άνοιγμα στις επιχειρήσεις και την καταπολέμηση διαφθοράς. Είναι ψηλά η Γεωργία. Διερωτώμε λοιπόν και ας διερωτηθούμε όλοι γιατί συζητούμε αυτό το θέμα σήμερα. Καλύτερα θα ήταν να βοηθούμε τη Γεωργία, να στηρίζουμε τις αρχές της Γεωργίας, τις προσπάθειες που καταβάλουν στη χώρα όσον αφορά στην προσπάθεια να την πλησιάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι αυτή είναι η Γεωργία που χρειαζόμαστε για μας σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα ας κοιτάξουμε εκ του σύνεγγυς τι κάνει η αντιπολίτευση. Ας δούμε κατά πόσο είναι προς όφελός της να έχει μια κυρίαρχη περήφανη χώρα ή μια χώρα που επηρεάζεται από τη Ρωσία. Τώρα και δίνω αμέσως το λόγο στο συνάδελφο κύριο Έλμαρ Μπροκ Νομίζω πως είναι απαραίτητο να βοηθήσουμε όλες αυτές τις χώρες της ανατολικής γειτονίας. Να τηρούνται οι ανάλογοι κανόνες για δημοκρατία, κράτος δικαίου, ελεύθερες εκλογές και όλα τα σχετικά. Βεβαίως ε, θα μπορέσουμε να τις ε, βοηθήσουμε για να φτάσουν αυτά τα οποία λέει το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο ΑΣΕ και βεβαίως μην ξεχνάτε πως ζήτησε η γεωργιανή κυβέρνηση να αποστηλουμε όσο δυνατόν περισσότερους παρατηρητές στις εκλογές. Θεωρώ πως είναι μια σχετικά καλή εξέλιξη. Κοιτάξτε, τώρα ένας χουλιγκάνος μπορεί να κάτσει 35 μέρες ε, εκλογές, 35 ε, μέρες με συγχωρείτε στη φυλακή, αλλού κάθε 7 χρόνια είναι διαφορά αυτή. Ε, επίσης, εάν σκεφτούμε πως υπάρχουν πάρα πολλοί τηλεοπτικοί σταθμοί με την ε, δυνατότητα του Κέρι το οποίο αποφασίστηκε από τις 27 ε, Ιουλίου και μετά θα ισχύσει, νομίζω πως είναι ικανοποιητική η κατάσταση. Επίσης, μην ξεχνάμε πως ε, ένα κόμμα μοιράζει τηλεοπτικούς δέκτες. Πράγματι, Μιλάτε για αδιαφάνεια. Ο άνθρωπος βεβαίως έχει κερδίσει 6 δισεκατομμύρια ευρώ στην ε, Ρωσία. Δεν ξέρω λοιπόν εάν όλα τα κόμματα τηρούν τους ίδιους κανόνες. Όταν βλέπουμε αποδείξεις πως αγοράζονται ψήφοι. Άλλα κόμματα έχουν 20 πλάσια από εσά στη διάθεσή τους από ό,τι κυβέρνηση. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι κάνει και η αντιπολίτευση εδώ πέρα, εάν είναι να μιλήσουμε για μια δίκαιη κρίση των ε, εκλογών. Επίσης δεν νομίζω πως η χρήση 18 εταιριών, αμερικανικών εταιριών συμβούλων ε, είναι και τόσο λιτότης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπρόκ. Ε, επόμενος ομιλητής είναι ο συνάδελφος κύριος Κρίστιαν Βιγγένιν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν νομίζω ότι τέτοιες συζητήσεις δημιουργούν ή δείχνουν τέτοιε συζητήσει Κανείς να αρνείται ότι η Γεωργία χρειαζονται αυτέ τις συζητησει κανεις να αρνειτε οτι η καλή σε πολλού τομεί. Αυτό είναι ενθαρρυντικό και υποδειγματική εξέλιξη. Τα μέλη του Κοινοβουλίου της Γεωργίας έπαιξαν πολύ ενεργό ε, και ενεργητικό ρόλο λοιπόν όσον αφορά την κοινοβουλευτική συνέλευση για τα ευρωπαϊκά θέματα τη οποία ε, προείδρευσα. Συμμετείχα μάλλον. Ε, λοιπόν, οι καλύτερε εταιρείε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι, οι εκλογέ δείχνουν πόσο βιώσιμη είναι μια δημοκρατία και πόσο όριμο είναι ένα πολιτικό σύστημα. Και ζητώ από του συναδέλφου να μην υπερβάλλουν, αλλά και να μην υποτιμούν τι πρόσφατε εξελίξει στη Γεωργία. Έχω την εντύπωση ότι και οι δύο πλευρέ χρησιμοποιούν τα όπλα στον πολιτικό πόλεμο που ακολουθεί. Από τη μία πλευρά, από την πλευρά του κόμματο τη ηγεσία, χρησιμοποιούνται οι διοικητικέ και νομικέ ε, δυνάμει που έχουν Απ' την άλλη πλευρά χρησιμοποιούν τους οικονομικούς ε, πόρους. Αν ακούσετε τις εξηγήσεις που δίνουν και δύο πλευρές για την κατάσταση στη Γεωργία, θα νομίζατε ότι αφορά δύο εντελώς διαφορετικές χώρες και αυτό ήδη είναι ένα σημάδι ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτή η κατάσταση πρέπει να σταματήσει και η πολιτική διαδικασία θα πρέπει να επανέλθει στην νομιμότητα. Ζητώ από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσουν όλη τη δύναμη που έχουν για να βοηθήσουν τη Γεωργία. Υπάρχουν διαθέσιμα μέσα διάφορα, τα ξέρετε καλύτερα, χρησιμοποιήστε τα τώρα. Διότι αν θέλετε να βοηθήσετε τη Γεωργία να διεξαγάγει δίκες και ελεύθερε εκλογές, η ώρα είναι τώρα ε, και όχι την ημέρα των εκλογών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βιγγέννη. Ε, δίνω τώρα το λόγο στον συνάδελφο κύριο Άνταμ Μπίλαν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν δούμε τη στάση του Κρεμλίνου έναντι της Γεωργίας, νομίζω ότι η δέσμευσή μας να κρατήσουμε τη Γεωργία στο δρόμο της, του οικονομικού μετασχηματισμού και της πολιτικής μεταρρύθμισης και της ελληνικής συμβίωσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ιδίω αυτό αφορά το νέο εκλογικό δίκαιο και το Σύνταγμα. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι η Ρωσία δεν θα παρέμβει σε όλα αυτά. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει ανάμειξή τους σε εσωτερικά θέματα όπως είναι η χρηματοδότηση των ομάδων αντιπολίτευσης. Ξέρουμε ότι η Γεωργία θέλει να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Εμείς είχαμε ζητήσει να υπάρξει μια συνέχεια των προσπαθειών για τη δημιουργία ενός χώρου ελευθέρων συναλλαγών και πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες της διαπραγματεύσης για μια εταιρική σχέση. Χρειάζεται επίσης να έχουμε και μια νέα πολιτική για τις ε, προξενικές θεωρήσεις για τις χώρες αυτές. Η Ρωσική Ομοσπονδία κατέχει ένα τμήμα του εδάφους <clears throat> της Γεωργίας και μάλιστα οργάνωσαν τον Οκτώβριο ή τον Σεπτέμβριο, τον Σεπτέμβριο μάλλον στρατιωτικές ασκήσεις όταν θα γίνουν και οι εκλογέ. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε ότι η Ρωσία θα αποσυρθεί από τα κατεχόμενα αυτά εδάφη. Ε, Mr. President, I have some... Κύριε Πρόεδρε, έχω κάποιες ανησυχίες για την κατάσταση στην Γεωργία και γύρω από τη Γεωργία. Υπάρχουν τρεις παράγοντες οι οποίοι συνδέονται με τις ε, εκλογές που μπορεί να οδηγήσουν σε αποσταθεροποίηση της γεωργίας και ακόμα να οδηγήσουν και σε νέες αιματηρές ε, παρεμβάσεις. Καταρχήν υπάρχουν τεράστια ποσά που έρχονται από τη Ρωσία για τη διαφθορά των πολιτικών και επίσης για την εξαγορά φτωχών με στόχο να μπορέσει να επανέλθει στο ρωσικό μαντρί η Γεωργία. Οι προσπάθειες του Γεωργιανού Κοινοβουλίου και της κυβέρνησης να αποφύγουν μια εκλογική εξατία η οποία θα είναι τελείως στρεβλή και απατηλού χαρακτήρα αντιμετωπίζονται από προπαγάνδα από την πλευρά του Κρεμλίνου που προσπαθούν να δώσουν την εντύπωση ότι υπάρχει περιορισμό τη ελευθερία. Δηλαδή θέλουν την ελευθερία να προωθούν ναζιστικού και φασιστικού χαρακτήρα επιθέσει εναντίον μη εθνοτικά γεωργιανών, μη ορθοδόξων γεωργιανών, αυτό που υποστηρίζουν τι μειονότητε κτλ. Δυστυχώ κάποια τέτοια κείμενα τα εκτιμούν ιδιαίτερα ορισμένοι Ευρωπαίοι φιλελεύθεροι, οι οποίοι δεν βλέπουν πέρα από τη μύτη τους. Ο στόχο είναι να κερδίσουν τα ρωσικά χρήματα. Ένα δεύτερος παράγον είναι οι ιδιαίτερα ισχυρές στρατιωτικές ασκήσεις που θα γίνουν λίγο πιο πέρα από τα, σύνορα της γεωργία και μπορεί να επηρεάσουν τις ε, διαμάχες εκεί. Τρίτος παράγον είναι η τωρινή ρωσική κάμψη στον οικονομικό τομέα και η κοινωνική κρίση η οποία προκύπτει με γεγονός ότι μπορεί να μην καταφέρει η άρχουσα τάξη να στρέψει τον, τον ρωσικό λαό εναντίον εξωτερικών υποτιθεμένων απα, ε, αντιπάλων. Χρειαζόμαστε λοιπόν τόλμη και θάρρος. Ε, επόμενος ομιλητής είναι ο συνάδελφος κύριος Ρίτσαρτ ε, Χάουιτ για Uh, Κύριε Πρόεδρε, οι ελεύθερες εκλογές ε, σημαίνουν και ελεύθερη προεκλογική εκστρατεία και σωστό είναι το ότι ε, θέτουμε εκ των προτέρων ζητήματα όπως η πρόσβαση στα ΜΜΕ, η βία κτλ. Και μάλιστα το να αποκλείουν από ορισμένα πακέτα συνδρομητικής τηλεόρασης στα κανάλια της αντιπολίτευσης πράγματι φαίνεται ε, παράδεκτο. Και επίσης βεβαίω έχουμε και την αντιμετώπιση του Gay Pride φέτος. Παρ' όλα αυτά, καλωσορίζει 400 παρατηρητές του ΟΑΣΕ η Γεωργία, έχει ένα διακομματικό όργανο που αποφασίζει για τις παραβιάσεις, παραβιάσεις και αντιλαμβάνομαι πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει την παρακολούθηση των ΜΜΕ, οπότε όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να ξέρουν πώς βλέπουμε Βεβαίως ε, τα ερωτήματά μας είναι σε ένα πνεύμα φιλίας ε, προς την χώρα και υπάρχει και το ζήτημα της ε, διοικητικής μεθοριακής γραμμής η οποία υφίσταται αυτή τη στιγμή και βεβαίως μην ξεχνάμε πως και Γεωργιανή αξιωματούχη η περσόνα non grata από κάποιες αρχές και βεβαίως να υπερυθμίσω πως μπλοκαρίστηκε η τροπολογία μου για να ε, γίνει λόγος για την παιδική εργασία ενώ η UNICEF έχει καταγγείλει ε, κάποια πράγματα. Αντιλαμβάνομαι πως κάποιοι θεωρούν πως προσπαθώ να βοηθήσω το κόμμα του κυρίου Σακασβίλη. Εμείς εδώ πέρα πρέπει να προωθήσουμε την δημοκρατία και δεν ε, το κάνουμε αυτό αν φαίνεται πως ελέγχουμε ένα κόμμα με διαφορετικό τρόπο από ό,τι ένα άλλο. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω στην αίθουσα τον κύριο Κυρίλοφ και ως εκ τούτου ανοίγει η διαδικασία Catch the Eye. Δίνω το λόγο στον κύριο Ντανζάν. Κύριε Πρόεδρε, το θέμα της ε, γεωργίας μας απασχολεί ιδιαίτερα. Υπήρξαν ε, επισκέψεις προσωπικότητων, υπάρχουν οι εκλογές τον Οκτώβριο, αλλά δεν είναι η πρώτη χώρα όπου γίνεται κάτι τέτοιο. Γνωρίζουμε πολύ καλά όμω γιατί μιλάμε σήμερα για τη γεωργία σήμερα. Μιλάμε για τη γεωργία γιατί κάποιο ολιγάρχη αποφάσισε να κατέβει στι εκλογέ δικαίωμά του και γιατί έχει πλημμυρίσει με δολάρια, ευρώ και ρούβλια τις εταιρείε ε, άσκησης πίεσης και λόμπι στην Ευρώπη, στο, στη Ουάσιγκτον και αλλού. Δεν μιλάμε σήμερα όμως για την παραβίαση των συμφωνιών ανακοχής από τη Ρωσία, ούτε για τη ρωσική κατοχή, ούτε για τις στρατιωτικές ασκήσεις που θα κάνουν οι Ρώσοι τον Οκτώβριο την εποχή των εκλογών, αλλά για να μιλήσουμε γενικά για την εκλογική διαδικασία στη Γεωργία. Υπενθυμίσατε ένα αριθμό ψηφισμάτων όπου εμείς τονίζουμε ότι πρέπει να είναι ανεξάρτητη η κοινωνία των πολιτών, να είναι ισχυρή και αξιόπιστη η κοινωνία των πολιτών. Δεν είναι τα εκατομμύρια ενό ολιγάρχη που κάνουν την κοινωνία των πολιτών ή την αντιπολίτευση ανεξάρτητη και αξιόπιστη. Δεν πρέπει να δώσουμε βέβαια επιταγή λευκό στον κύριο Σακιασβήρη αλλά ούτε και σε αυτόν τον νεόφερτο ολιγάρχη, ο οποίος μου φαίνεται ακόμα πιο επικίνδυνος. Επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Όγιουλαντ. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι εκλογέ είναι δύσκολη εποχή σε οποιαδήποτε δημοκρατική χώρα, οπότε συμμερίζομαι την άποψη κάποιων συναδέλφων που παρεξηγούν γιατί διεξάγεται αυτή η συζήτηση τώρα και γιατί είναι στην ημερήσια διάταξη. Όμω, Πραγματικά ελεύθερες και δίκαιες εκλογές δεν αφορούν μόνο το σεβασμό των διατάξεων του νόμου και το πνεύμα της εκλογικής διαδικασίας και των αποτελεσμάτων. Επίσης αφορούν και το θεμητό ανταγωνισμό, τον τίμιο ανταγωνισμό και να μην γίνονται ε, λόγοι, γίνονται λόγοι που δημιουργούν μισαλλοδοξία. Ελπίζουμε ότι όσοι δυνάμεις στη Γεωργία θα δείξουν αυτοσυγκράτηση και δεν θα φτάσουν να οδηγήσουν την πολιτική στους δρόμους, κάτι που οδηγήσει σε βίες συγκρούσεις. Επιπλέον ο ρωσικός στρατός είτε κάνουν ε, έχοντας, κάνοντας ασκή στην περιοχή και ένα κομμάτι της χώρας να κατέχεται από τις ρωσικές δυνάμεις αυτή την εποχή. Αυτό ισχύει. Είναι μια νέα δημοκρατία η Γεωργία που χρειάζεται υποστήριξη στις προσπάθειές της να ενταχθεί περισσότερο στους διάφορους θεσμούς, τους διατλαντικούς και τους ευρωπαϊκούς. Πρέπει να βοηθήσουμε την κυβέρνηση να συνεχίσει τις τρέχουσες μεταρρυθμίσεις διαβεβαιώντας και καθησυχάζοντας τη Γεωργία για τις προοπτικές που έχει. Ελπίζουμε ότι η παγίωση της δημοκρατίας Χρειάζεται τη βοήθειά μας και χρειάζεται και σταθερή συνεργασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενος ομιλητής είναι ο συνάδελφος κύριος Τάνοκ. Ο πρόεδρος Σακασβίλη ε, είναι βεβαίως μεγάλος πολιτικός επιζών παρά το ότι έχασε δύο επαρχίε ε, μετά τον πόλεμο με την Ρωσία. Κατάφερε να φέρει τη χώρα του πιο κοντά στην Ευρώπη με τις διάφορες συμφωνίες σύνδεσης και στο ΝΑΤΟ και έχει καταπολεμήσει τη διαφθορά και ενισχύει την ελεύθερη οικονομία. Έχει ορίσει τον πεπειραμένο Μεραπισβήλη ως Πρωθυπουργό, ο οποίος πρέπει τώρα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, αλλά ελπίζω να υπάρξουν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ του δισεκατομμυριούχου Ιμπανισβήλη, του ε, ονείρου για την γεωργία και της ε, κυβέρνησης. Η δημοκρατία είναι κάτι το οποίο κερδίζεται δύσκολα και πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή τη μικρή χώρα του Καυκάσου. Ελπίζω επίσης να υπάρξει μακροπρόθεσμη αποστολή παρατηρητών της Ένωσης για να έχουμε ελεύθερες εκλογές στην όμορφη αυτή η χώρα. Το λόγο έχει τώρα ο συνάδελφος κύριος Κέλαμ. Ευχαριστώ πολύ. Οι εκλογές του Οκτωβρίου σίγουρα θα αποτελέσουν δοκιμή για τη δημοκρατική πρόοδο της Γεωργίας και κατά κάποιο τρόπο θα είναι και μια δοκιμή για τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ενώσης όσον αφορά αυτή τη χώρα. Τώρα που πλησίασε πράγμα την Ευρωπαϊκή Ένωση η Γεωργία, θα ήταν αφελές να αναμένουμε ότι δεν θα υπάρχουν εξωτερικές επιρροές προσπαθώντας να αλλάξουν την πορεία της Γεωργίας, να την απομακρύνουν από τον ευρωπαϊκό δρόμο λαϊκιστικές και εθνικιστικές δυνάμεις αναδύονται. Και αυτό δημιουργεί σωστά ανησυχίες. Ο γέντης, ο κ. Ιβανισβίλη αυτών των δυνάμεων, είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος και στη Λουκόελ και στην Κάσπρομ. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα για να ξέρουμε με ποιανού νου το μέρος είναι. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να επιμείνει να ισχύσει η συμφωνία της Μόσχας και να επιμείνει να επιτραπεί σε παρατητές Ευρωπαϊκής Ενώσεως να επιβλέπουν την κατεχόμενη περιοχή. Αυτή θα είναι μια κίνηση που θα δείχνει την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην περιοχή. Ευχαριστώ. Κύριε Κέλλαμ, ε, τελευταίος ομιλητής, ο συνάδελφος κύριος Μάγερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε είναι ένας πολύ σημαντικός και στρατηγικά σημαντικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, περιοχή του Καυκάσου και φυσικά έχουμε και ιστορικούς και θρησκευτικούς ε, θεσμούς, ε, δεσμούς με τη χώρα αυτή. Έχουμε μεγάλες διαδηλώσεις κατά του κ. Σακιασβίλη, 80.000 διαδήλωσαν πρόσφατα. Υπάρχει το θέμα της, των, των πολιτικών και ατομικών δικαιωμάτων τα οποία έχουν περιοριστεί κατά τη διάρκεια της θητείας του κυρίου Σακιασβίλη. Και έχουμε το, την απειλή του γείτονα από, το, από την ρωσική πλευρά που απειλεί την νεαρή δημοκρατία της Γεωργίας. Η Γεωργία είναι τμήμα της ε, ομάδος χωρών που βρίσκονται στην πολιτεία, στην, στην Ευρωπαϊκή Ανατολική Συμμαχία. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι οι δημοκρατικές αρχές δεν θα χαθούν στη Γεωργία και θα κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και υπάτης εκπροσώπου για τις εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική ασφάλεια, το λόγο έχει ο Πρόεδρος κ. Μαυρογέννης Ανδρέας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. I sincerely thank all... Ευχαριστώ ειλικρινώς όλους τους βουλευτές που τοποθετήθηκαν για αυτό το σημαντικό θέμα. Ξεκινήσω με μια γενική δήλωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποδέχεται την εργαλειοποίηση της δημοκρατικής διαδικασίας για σκοπούς απότερους ή για να πλαστογραφηθεί η Λαϊκή Βούληση από οποιονδήποτε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί πως ε, πρέπει να πιστεύει στις ε, ελεύθερες και δίκαιες εκλογές και πως ε, ο δίκαιος ανταγωνισμός των κομμάτων και η σωστή συμμετοχή στις εκλογές έχουν θεμελιώδη σημασία για τα αποτελέσματα αυτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει πως οι πολιτικές διώξεις, με άμεσες ή έμεσες, με οποιονδήποτε τρόπο, είτε μιλάμε για επιλεκτική χρήση της δικαιοσύνης, δεν είναι συμβατές με τις δημοκρατικές αξίες. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί και θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση στην Γεωργία μέχρι τις εκλογές αλλά και την διεξαγωγή των εκλογών. Η κυρία Άστον είπε εκπρόσωπο ε, συνάντησε την προηγούμενη εβδομάδα τον πρόεδρο Σάκασβιλ. Οι υπηρεσίε τη ε, συναντήθηκαν με εκπροσώπου του συνασπισμού του Ονείρου για τη Γεωργία και οι δύο πλευρέ ζήτησαν μεγαλύτερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ήδη κάνει πολλά σε συνεργασία με τον ΟΑΣΕ και όσον αφορά την παρακολούθηση των ΜΜΕ. Κάτι στο οποίο αναφερθήκατε πολλοί από εσά. Όμως, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης επίσης εξετάζει το πώς μπορεί να στηρίξει περισσότερο την διαδικασία για να επιτευχθεί μέγιστη διαφάνεια. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της ε, παρα... πάνω παρακολούθησης ε, της διεξαγωγής των εκλογών, exit poll και της ε, στήριξης από τους διεθνείς οργανισμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συστήσει μια ειδική ομάδα δράσης με επικεφαλή στην αντιπροσωπεία επιτόπου. Οπότε παρακολουθούμε και βοηθούμε. Γενικά η θέση μας είναι σαφής για την Γεωργία. Είμαστε υπέρ των στενών σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε δει ε, αρκετά καλή πρόοδο στα θέματα της ε, ανατολικής ε, εταιρικής σχέσης και προχωρούμε επίσης προς την κατεύθυνση της απελευθέρωσης της βίζας. Υπάρχουν και άλλα στρατηγικά συμφέροντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει την αυξανόμενη σημασία της Γεωργίας ως μια χώρα διαμετακόμισης ε, ενέργειας και ιδιαίτερα όσον αφορά τον νότιο ενεργειακό διάδρομο και αναγνωρίζουμε την σημαντική συνεισφορά της στις ειρηνευτικές προσπάθειες ανά την Ιφίλιο. Έχουμε δει πολλές θετικέ αλλαγές από την από την επανάσταση των τριαντάφυλων. Και βεβαίω αναμένουμε ακόμα τα αριθμιστικέ προσπάθειε ειδικά στην τομέα τη δικαιοσύνη στην οικονομία και την κοινωνική ε, ζωή και βεβαίω και τι περιθωριοποιημένε ομάδε. Αλλά πάνω απ' όλα η περιφερειακή ασφάλεια και οι δημοκρατικές εξελίξεις είναι τα σημεία κλειδιά για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν πλήρω τα ωφέλη της Συμφωνίας Σύνδεσης. Ευχαριστώ. Προεδρία και κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση έληξε. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι δήλωση Αντιπροέδρου της Επιτροπής, πάτηση εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Θέμα η κατάσταση στην Συρία. Ο κύριος Ανδρέας Μαυρογιάννης, εκπρόσωπος Προεδρίας, έχει το λόγο εξ ονόματος της Αντιπροέδρου